Ladies and gentlemen, good afternoon. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα. Welcome to this extraordinary meeting Καλώς ήρθατε σε αυτήν την εξαιρετική συνάντηση της Επιτροπής μας. Έχουμε δύο ψηφοφορίες στη μέση διάταξη σήμερα. Ελπίζω όλοι να έχετε βάλει τις κάρτες σας στο κατάλληλο σημείο διότι και οι δύο ψηφοφορίες ε, θα γίνουν με κάρτα Ξεκινούμε με την οδηγία για το copyright. Άρχεται η ψηφοφορία. Ε, we have one e ε, ψηφίζει ένας παραπάνω από το ΕΛΚ. Τώρα, τώρα που καταστάθηκε η τάξη, πέρας ψηφοφορίας Ευρεία πλειοψηφία υπέρ. to the Συγχαρητήρια στον εισηγητή και τους κοιόδης εισηγητές, βεβαίως, προφανώς. Και τώρα πάμε στην δεύτερη ψηφοφορία για το, ε, το ε, πιστοποιητικό προστασίας για τα ιατρικά προϊόντα. Έχει την ψηφοφορία. Πάλι περισσεύει κάποιος από το ΕΛΚ. Εξακολουθεί να υπάρχει υπεράριθμος στο ΕΛΚ. Πέρας ψηφοφορίας. Δεν μπορώ να το πράξω όμως αυτό, διότι εξακολουθούμε να έχουμε ένα μέρος του ΕΛΚ που περισσεύει. Α, τώρα, τώρα είμαστε εντάξει. Πολύ ωραία, εγκρίνεται με ευρεία πλειοψηφία συγχαρητήρια στον εισηγητή και στους κοιόδης εισηγητές. And thank you for attending this... Και σας ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ.